Καλημέρα σε όλους. Να σας ενημερώσω για κάτι ξεκινώντας. Θα πρέπει το σημείο 10 George Lyon θα πρέπει να το πάμε το απόγευμα για την καλλιέργεια γενετικά τροπομένων οργανισμών και να έχουμε έτσι όλους τους εμπειρογνώμονες, τους επίσημους που έχουμε προσκαλέσει για την καλλιέργεια αυτών γενικά τροπομένων οργανισμών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν ε, και τώρα για τα κράτη-μέλη πώς θα μπορούσαν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια παρόμοιων οργανισμών θα πάει το απόγευμα στις 5. Τα υπόλοιπα όλα παραμένουν στη θέση τους. Ξεκινάμε λοιπόν και Ελπίζω να έχετε όλη την κάρτα για την ψηφοφορία σας. Ξεκινάμε το σημείο 8. Αναγνώριση της γεωργίας σαν ένα στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επισητιστικής ασφάλειας. Η συγήτριά μας είναι η Ντατσιάνα Οκτάβια Σάρμπου. Έχει το λόγο. Έχουμε 185 τροπολογίες στην πρωτοβουλία αυτή, αλλά ε, οι συγητή και οι σκιώδεις συγητέ εργάστηκαν σκληρά και έτσι πέτυχαν συμβαστικέ τροπολογίε. Ελπίζω ότι πολύ πολύ γρήγορα θα φτάσουμε και στην ψηφοφορία. Η εισηγήτρια Ντατσάνα Σάρμπου έχει το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, δεν ε, θα επεκταθώ γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την υποστήριξή της και επίσης θα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους χιώδης συγητές και όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή γιατί ιδιαίτερα με βοήθησαν για την επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Πολύ καλά λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Ντατσάνα Οκτάβια Σάρμπου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία μας. Ξεκινάμε με τη συμβαστική λύση πρόταση 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πρέπει να λάβω το λόγο. Ναι, ζήτησε το λόγο. Ή όχι. Ναι. Α, για πρώτη φορά σήμερα δεν έχω την κάρτα μαζί μου. Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να ψηφίσω έτσι για ανατάσσος χειρός. Ξέχασε την κάρτα μου. Ε, ο πρόεδρος. Εντάξει, το σημειώνουμε. Ξεκινούμε λοιπόν τη ε, ψηφοφορία Συμβαστική Λύση 1, πρόταση 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ και αν ψήφισαν όλοι. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισε και ο Μάρκ. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, περνάει. Τροπολογία 6. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 6. Πέρας ψηφοφορίας για την 6. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 7 τώρα. Ψηφίζουμε πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 8. Και αν ψήφισαν όλοι. Πέρας και απορρίπτεται. Η 9 τώρα. Τροπολογία 9 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η εννέα. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε για την 11. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας για την 11. Απορρίπτεται με μία ψήφο περισσότερη ε, το όχι. 12. Ψηφίζουμε για την 12 τώρα. Και αν ψήφισαν όλοι, τότε πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψηφίζουμε. 14. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ για τη 15. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 15. 16 τώρα. Ψηφίζουμε για την 16. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 17. Ψηφίζουμε για το 17. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17. 19 τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας για το 19. Εγκρίνεται. 18. Λούλιν. Ψηφίζουμε για το 18. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Όχι. Ή ναι, ναι. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε για την 20. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 22 έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μαγκίνες ε, στην οθόνη ε, εμφανίζονται τα αποτελέσματα τριών ψηφοφοριών πίσω και μας μπερδεύει. Δηλαδή βλέπουμε κάτι και ακούμε κάτι άλλο. Θα ήταν καλό να φαίνονται αυτά τα οποία λέτε στην οθόνη. Εντάξει, ευχαριστούμε την κυρία Μαγκίνες. Θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Τροπολογία 22. Ψηφίζουμε για την 22. Να δούμε αν μπορούμε να συγχρονίσουμε το αποτέλεσμα με το που φαίνεται με αυτό που αναγγέλλεται. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μαγκίνες, αυτός ο αριθμός για το 17 είναι ο αριθμός ψηφοφορίας. Δεν έχει σχέση με, τον, ε, με την την ίδια, με τον ίδιο το αριθμό της τροπολογίας. Είναι 17η ψηφοφορία, όχι η τροπολογία 17. Λοιπόν, ακούστε τον πρόεδρό σας, μην μην κοιτάζετε την οθόνη. Ψηφίσαμε. Γκίνες λοιπόν. Ψηφίζουμε για την 23. Πέρας ψηφοφορίας για την 23. Εγκρίνεται. 24. Ψηφίζουμε για την 24. 24. Εγκρίνεται. 25. Ψηφίζουμε για την 25. απορρίπτεται. 28 Μα γινες. 28 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 29 ψηφίζουμε και την 29. Ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 29. Η 30 τώρα. Ψηφίζουμε για την 30. Πέρα ψηφοφορίες. Εγκρίνεται η 30. Η 31 τώρα. Όσλιν. 31 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 36 Λάιον και άλλοι και οι υπόλοιποι ψηφίζουμε για την 36. 36. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε, επαναλαμβάνω. Εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία 37. Ψηφίζουμε για 37. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Ψηφίζουμε για 39. 39 λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όχι, όχι. Ίσα ίσα. 18-18 το αποτέλεσμα. Ο Άλμπερτ όμως δεν έχει την κάρτα του. 40 ταραμπέλα. Το πρώτο μέρος της 40. Πρώτο μέρος της 40. 40. Πρώτο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 ταραμπέλα, αλλά το δεύτερο μέρος τώρα. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο μέρος. Πάμε στη 41. Ψηφίζουμε. 41. 41. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 41. 42. Ψηφίζουμε. 42. Πέρας. Εγκρίνεται η 42. Συμβαστική πρόταση 14. Ψηφίζουμε. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 14. Και τώρα η 44. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 45. Ψηφίζουμε για τη 45. Πέρας. Απορρίπτεται η 45. 46. Ψηφίζουμε για τη 46. Πέρας. Εγκρίνεται η 46. 48. Ashworth. Ψηφίζουμε για τη 48. Πέρας. Απορρίπτεται η 48. 49. Ψηφίζουμε για τη 49. Πέρας. Απορρίπτεται η 49. 50. Ψηφίζουμε για την 50. Γέγκλη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 52. Όχι. Η 50. 51. Ψηφίζουμε για την 51. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Έλβορτ, Λάιον και άλλοι. Ψηφίζουμε για την 52. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε. 16. Πέρας. Εγκρίνεται η 16. 66 ψηφίζουμε. 66 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 4. Μισό λεπτό να πάρουμε και το καφεδάκι μας. Διάλειμμα. Απορρίπτεται φωνάζει κάποιο. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη συμβαστική 4. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε ήδη αυτή. Πάμε στην 5 τότε, συμβαστική 5. Πέρασε ψηφορίες. Εγκρίνεται. Μαγκίνες 76. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα 80 Ashworth. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 80. 81. Ψηφίζουμε για την 81. Πέρας. Εγκρίνεται 81. 82. Ψηφίζουμε. 82. Πέρας εγκρίνεται. 83. Ψηφίζουμε για την 83. 83. Πέρας εγκρίνεται 84 πέρας εγκρίνεται 84 συμβαστική πρόταση 6 ψηφίζουμε την 6 πέρας εγκρίνεται 88. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 τώρα. Ψηφίζουμε για την 89. Πέρας. Εγκρίνεται 89. 90. Ψηφίζουμε για την 90. Πέρας. Εγκρίνεται η 90. Ε, ο Άλμπερτ καταψήφισε. Με ενδιαφέρον αυτό. 91. Ψηφίζουμε την 91. Πέρας. Απορρίπτεται. 92. Ψηφίζουμε για την 92. Πέρας. Εγκρίνεται. 93. Ψηφίζουμε 93. Πέρας. Εγκρίνεται. 94. Ψηφίζουμε για την 94. Πέρας. Απορρίπτεται. 95. Ψηφίζουμε για την 95. Πέρας. Απορρίπτεται. 96. Ντάνσιδα. 96. Πέρας. Απορρίπτεται. 97. Ψηφίζουμε για την 97. Πέρας. Απορρίπτεται 97. 98. Ψηφίζουμε για την 98. Πέρας. Απορρίπτεται. 100. Ψηφίζουμε την 100. Πέρας. Απορρίπτεται η 100. 99. 99. Ψηφίζουμε την 99. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 99. Ψηφίζουμε την 102 Ashworth. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 92. 103. Γκρατφέλντερ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 103. Συμβαστική λύση 12. Πρόταση 12. Συμβαστική πρόταση 12. Πέρα, ε, ψηφίζουμε. Τε, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7. Ψηφίζουμε για την 7. Πέρας. Εγκρίνεται η συμβαστική 7. Συμβαστική πρόταση 8. Ψηφίζουμε για την 8. πέρασε Εγκρίνεται η 8. Πάμε στην 118 τώρα. λίγο κι άλλο. Ψηφίζουμε την 118. πέρασε Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 117 Γέγκερ. Ψηφίζουμε για την 117. Πέρας. Εγκρίνεται 117. 122. Ψηφίζουμε την 122. Πέρας. Εγκρίνεται η 122. 123. Ψηφίζουμε για την 123. Πέρας. Εγκρίνεται η 123. 124. Ψηφίζουμε για την 124. Πέρας. Απορρίπτεται η 124. 125. Ψηφίζουμε για την 125. Πέρας. Απορρίπτεται η 125. 126 ψηφίζουμε για την 126 εγκρίνεται 126 128 Νικολέσκου ψηφίζουμε για την 128 πέρας εγκρίνεται η 128 127 τώρα ψηφίζουμε για την 127 εγκρίνεται 127 Συμβαστική πρόταση 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 135. Ψηφίζουμε για την 135. Πέρας. Εγκρίνεται 135. 136. Ψηφίζουμε για την 136. Πέρας. Εγκρίνεται 136. 140. Ψηφίζουμε για την 140. Πέρας. Εγκρίνεται 140. Συμβαστική πρόταση 15. Ψηφίζουμε για την 15. Πέρασε. Εγκρίνεται 115. Και τώρα 145. Ντάνσιδα. Πέρας. Εγκρίνεται 145. 146 σκοτά. Ψηφίζουμε την 146. Πέρας. Εγκρίνεται 146. 147. Ψηφίζουμε για την, 147. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση 9. 9. Ψηφίζουμε για την 9. Πέρας Εγκρίνεται η συμβαστική εννέα. 157. Ψηφίζουμε για την 157. Πέρας. Απορρίπτεται 157. 159. Νεγκολέσκο. Ψηφίζουμε για την 159. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική πρόταση 10 σε δύο ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο μέρος της 10. Πρώτο μέρος. Πέρας. Εγκρίνεται. πάντα τη συμβαστική 10, αλλά το δεύτερο μέρος ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Μπερδεύομαι, μπερδεύομαι. Το δεύτερο μέρος απορρίπτεται της 10 της συμβαστικής. 171 Νικουλέσκου ψηφίζουμε την 100, για την 171 πέρας απορρίπτεται 171 173 ψηφίζουμε για την 173 πέρας απορρίπτεται η 173 174 Παπαστάμκου και άλλων. Ψηφίζουμε για την 174. Πέρασε. Εγκρίνεται 174. 180 τώρα, Ντάντεμ Κύπο. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 180 Πέρας. Απορρίπτεται 180. 181 μαγκίνες. Ψηφίζουμε 181. Εγκρίνεται 181. Τι θα ψηφίσουμε τώρα από τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Απορρίπτεται η δύο. Η τρία. Ψηφίζουμε για την τρία της περιβάλλοντος. Ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται η 3. Τροπολογία 4. Όχι. 7. Πάμε στην 7. Ψηφίζουμε για την 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πέρας. Απορρίπτεται η 7. Η 8 τώρα. Τις απορρίπτουμε όλες λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, 8. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 8. Τροπολογία 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 9. 10. Ψηφίζουμε για τη 10. Πέρας. Απορρίπτεται η 10. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε για την 11. Πέρας. Εγκρίνεται η 11. 14. Ψηφίζουμε για την 14. Πέρας. Εγκρίνεται η 14. 16 τώρα. Ψηφίζουμε για τη 16. Πέρας. Εγκρίνεται η 16. 17. Ψηφίζουμε για 17. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Ψηφίζουμε για τη 18. Πέρας. Απορρίπτεται η 18. 20. Ψηφίζουμε για την 20. Πέρας. Εγκρίνεται η 20. 21. Ψηφίζουμε για την 21. Πέρας. Απορρίπτεται 21. 22. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 20. 23 ε. τώρα. Ψηφίζουμε για την 23. Το ίδιο. Απορρίπτεται 23. 24. Ψηφίζουμε για την 24. Απορρίπτεται 24. 26. Ψηφίζουμε για την 26. Πέρας. Απορρίπτεται 26. 27. Ψηφίζουμε για την 27. Απορρίπτεται 27. 29. Ψηφίζουμε για την 29. Εγκρίνεται 29. 33. Ψηφίζουμε για 33. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Ψηφίζουμε για 34. Απορρίπτεται. 35. Ψηφίζουμε για 35. Απορρίπτεται και η 35. Αυτά. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση τροποποιημένη. Ψηφίζουμε. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και συγχαρτήρια στην εισηγητριά μας την κυρία Σάρμπου. ξεκουραστείτε λίγο και ξαναξεκινάμε με την ψηφοφορία. Συνάδελφοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία μας. Είναι η πράσινη βίβλος της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμασία των δασών εν ώψη της κλιματικής αλλαγής. Συντάκτης γνωμοδότησης, ο Αντιπρόεδρος Νισκουλέσκου. 112 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Και οι συγητές και οι συγητές έκλεισαν και συμβαστικές ε, προτάσεις ε, που κάνουν να συγκλίνουν οι απόψεις επιτροπής μας. Και συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι σημερινές τροπολογίες όπως θα εγκριθούν θα ενταχθούν στην τελική έκθεση. Τώρα εισηγητής Νικουλέσκου. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υπέβαλαν τροπολογίες και ιδιαίτερα τον σκιώδη εισηγητή για το ανοιχτό τους πνεύμα στις ε, διαβουλεύσεις Πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπημένες αυτές οι συμβιβαστικές τροπολογίες και ότι αντανακλούν τις απόψεις της Επιτροπής μας. Και ευχαριστώ επίσης ε, τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Νικουλέσκου και ξεκινάμε με τις ε, ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε την συμβαστική 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ την 1. για... Μήπως κάποιος μπορεί να μας πει κάτι τι γίνεται για την ομάδα των σουλιστών. Ναι. Εντάξει, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε για την 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε για τη 10. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Ψηφίζουμε για την 11. Ψηφίζουμε για την 11. Πέρας. Απορρίπτεται η 11. 12. Ψηφίζουμε για τη 12. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Ψηφίζουμε για 13. Πέρας. Εγκρίνεται. Dichiaro aperta la votazione sul 16. Votazione sul... Ψηφίζουμε για 16. Πέρας. Εγκρίνεται η 16. 17. Ψηφίζουμε για 17. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα η 19. Ψηφίζουμε για την 19. 19. Πέρας. Εγκρίνεται 19. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε για την 20. Εγκρίνεται. 20. 21 τώρα. Ψηφίζουμε για την 21. Πέρας, εγκρίνεται 21. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 3. Τροπολογία 30. Τροπολογία 30 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Πέρας. Απορρίπτεται. 33 τώρα. 33. Ψηφίζουμε και 33. Πέρας απορρίπτεται. 34. Ψηφίζουμε, πέρας, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 4. 4 λοιπόν. Ψηφίζουμε, πέρας, εγκρίνεται η 4. Τροπολογία 43. Ψηφίζουμε για τη 43. Πέρας. Εγκρίνεται η 43. 45. Ψηφίζουμε πέρας. 46. Απορρίπτεται η προηγούμενη. 46. Και αν ψήφισαν όλοι. 46. Απορρίπτεται. 47 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 48. Ψηφίζουμε τη 48. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. 50. Η 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Συμβιβαστική 5. Συμβιβαστική 5. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. 57. Ένα λεπτό λέει ο πρόεδρος. Να επαναλάβουμε την τροπολογία 57. 57. Ψηφίζουμε ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Άρχεται ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 67. Α, Ψηφίζουμε την 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 74. Τροπολογία 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε απορρίπτεται. 75 75 Άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται. 76 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 77. Άρχεται η ψηφοφορία. 77. Απορρίπτεται. 78. Ψηφίσατε όλη την 78. Εγκρίνεται. 79. Ψηφίσατε όλη την 79. Έκλεισε, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρο, ε, ε, εγκρίνεται. Η 83, 83. Άρχεται η ψηφοφορία για την 83. Έληξε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 8. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σημειβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Σημειβαστική 11. Εγκρίνεται. 107. Ε, ε, Τροπολογία 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 107. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προτείνουμε την πρόταση ως τροποποιησίσα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Συγχαρητήρια. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Νικουλέσκου για την υπερψήφιση. Λοιπόν, συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα ακόμα θέμα στην μερίσια διάταξη. Το τελευταίο του πρωινού. Όπως σας είπα, στην αρχή της συνεδρίασης, το σημείο 10 για τα γενετικά τροποποιημένα θα συζητηθεί στις 5 με τους εμπειρογνώμονες. Οπότε μας ε, απομένει μόνο το σημείο 11 το πρωί, γεωργία και διεθνές εμπόριο. Ο κύριος Παπαστάμκος είναι ήδη εδώ και σας υπενθυμίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι οι διεθνείς συμφωνίες για το εμπόριο και η απελευθέρωση του εμπορίου σε αγροτικά προϊόντα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας παρακαλώ να παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό, το οποίο έχει επιπτώσει στην ποιότητα, <clears throat> στην ανταγωνιστικότητα και κοινωνικές επιπτώσεις. Στο μέλλον πρέπει να μειώσουμε ρίζικα τις τρευλώσεις στην αγορά αυτή που δημιουργείται από εμπορευόμενους του κλάδου που δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που χαίρονται ε, άνομων ε, πλέον εκτιμάτων ε, παραβιάζοντας τους κανονισμούς μας. Πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Παπαστάμκο για την εξαιρετική του εργασία. Επίσης, Έχουμε την κυρία Κρίστα από την Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου η οποία είναι η συνδεδεμένη επιτροπή βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού που θα, μας, που θα συμβάλλει στη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Γιώργο. Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις οι οποίες ε, αναδεικνύουν ε, και την σπουδαιότητα ε, της θεματικής της εν λόγω έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει. Ο συνολικός αριθμός τροπολογιών ανέρχεται σε 127. Θεωρώ ότι υπάρχει σύγκληση στα κύρια σημεία της έκθεσης και όπως είναι φυσικό θα προτείνω ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες και συγχωνεύσεις τροπολογιών προκειμένου να υπάρξει συνοχή στο κείμενο της έκθεσης αλλά και ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες εισάγουν νέα σημεία στο κείμενο της έκθεσης τις οποίες και στηρίζω. Οι τροπολογίες τις οποίες θα αναφέρω ευθύ αμέσω στις οποίε θα αναφερθώ κατωτέρω είναι τροπολογίες τις οποίε ανεπιφύλακτα τις στηρίζω. Στηρίζω λοιπόν τι τροπολογίε με τι οποίε υπογραμμίζεται η ανάγκη παροχή αποζημιώσεων στους γεωργού της ΕΕ οι οποίοι πλήττονται από τι εμπορικέ συμφωνίε με τρίτε χώρες. Επίσης τροπολογία που αναφέρεται στι επιπτώσει των εμπορικών συμφωνιών στις απόκεντρες περιοχές, στα ε, outermost regions, εκεί οι τροπολογίες όπου, σύμφωνα με τι οποίε καλείται η Κομισιόν να προβεί στις αναγκαίε μεταρρυθμίσει για τη βελτίωση του συστήματος τιμών εισόδου για τα οποροκυπευτικά, για την ανάδειξη προβληματικών πτυχών της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο, η τροπολογία που αναφέρει τις ανησυχίες για τη συμφωνία σχετικά με τις μπανάνες, για την πρόταση της Επιτροπής για τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν, εν είδη με τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, εν προκειμένου δε στον τομέα της ε, βιοεθανόλης, ένα θέμα το οποίο συζητείται σήμερα και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, στην Ίντα, τροπολογίες που αναφέρονται στην διασφάλιση συμμετρικών συμμετρών, συμμετρικών παραχωρήσεων στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ε, στα FTAs με χώρες οι οποίες διαθέτουν σημαντική παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα στον τομέα της γεωργίας. Υπογραμμίζω τις δύο τροπολογίες τις οποίες καταθέσαμε από κοινού 16 συνάδελφοι ε, σχετικά με τα συστατικά στα προϊόντα καπνού ε, τροπολογίες με τις οποίες ενθαρρύνεται η Επιτροπή η Κομισιόν να προβεί σε ενεργό χρήση των εργαλείων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των μη δικαιολογημένων εμπορικών φραγμών, εμπορικών εμποδίων που επιβάλλουν τρίτες χώρες στις εξαγωγές προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης αυτές που, με τις οποίες επισημαίνονται τα θετικά στοιχεία της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοτιού Κορέας και εκεί όπου ζητείται η πληροφόρηση και εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. ένα θέμα στο οποίο μας το έχει φωτίσει όλος ιδιαίτερος η συνάδελφος η κυρία Γέγλε αυτό το θέμα Επίσης θεωρώ ότι ένα ιδιαίτερος κρίσιμο ζήτημα για την δική μας Επιτροπή είναι τα πρότυπα και οι προδιαγραφές των εργαζομένων στην ΕΕ, των εισαγωμένων συγγνώμη, στην ΕΕ προϊόντων. Στο σχέδιο της έκθεσής μου κάνω λόγο για ισοδύναμες, για αντίστοιχες equivalent προδιαγραφές συμμόρφωσης. Ορισμένοι συνάδελφοι ζητούν με τις τροπολογίες τους την επιβολή ίσων, ιδίων, equal, same απαιτήσεων στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της ε, ευζοίας των ζώων, στο animal welfare και σε άλλα. Ε, πιστεύω ότι ο, ο, ο καλύτερος όρος, ο προτιμότερος όρος είναι το ισοδύναμες, το αντίστοιχες και όχι το same ε, ή το equal δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα. Θα προτείνω επίσης κάποια διατύπωση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Τέλος, θα ήθελα να επιθυμίσω, το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι εφαρμόζεται η κατάρθρον 50 ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της δικής μας Επιτροπής, της Επιτροπής Άγκρη και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της ΙΝΤΑ. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ της κυρίας Γκβίστχουτ τίθε σήμερα το μεσημέρι σε ψηφοφορία. Ε, θα λάβουμε υπόψη ασφαλώς και θα εσωματώσουμε τα σημεία αρμοδιότητας της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε και θα, τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω τις δημιουργικές συνεισφορές των συναδέλφων σε αυτή την έκθεση που κατατέθηκαν με τις πάρα πολύ γόνιμες ε, τροπολογίες τους και σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό οι τροπολογίες αυτές θα είναι αποτυπωμένες και στο τελικό κείμενο ε, της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Γιώργο για την εξαιρετική σου εργασία. Και την κυρία Κουιστάουτ περιμένουμε, δεν ήρθε ακόμα. Λοιπόν, ε, περιμένουμε την εισηγήτριά μας η γνωμοδότηση ε, από το Διεθνές Εμπόριο. Περιμένοντάς την λοιπόν, ξεκινάμε την όλη συζήτηση. Ε, ήδη μας ενημέρωσε ο κύριος και ο κύριος Μάτο έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρο. Σύντομα, σύντομα να συγχαρώ τον κύριο Παπαστάμκο. Νομίζω ότι συνέταξε μια καλή έκθεση που δεν ήταν εύκολη. Θα έπρεπε να συγκλίνουν αρκετά σημεία, τα κατάφερε και ανάμεσα σε αυτά και το δικό μου σημείο. Άρχισε κριτική ιδιαίτερη για το ελεύθερο εμπόριο πολλές φορές γιατί το, κόστο αυτός, το κόστος αυτός των ε, συμφωνιών θα βαρύνει σε ορισμένο τομέα ε, τον γεωργικό ιδιαίτερα. Και γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να γίνουν πολλά, πολλά να καταφέρει σε αυτό. Και υπήρχε και ένα βασικό πρόβλημα, το είπα από πάντα, ότι δεν γίνονται σωστέ διαπραγματεύσει. Αν δεν γίνουν σωστέ διαπραγματεύσει, τότε αρχίζουν να αντισταθμίσει από εδώ και από εκεί. Καλύτερη διαπραγμάτευση, λιγότερε παραχωρήσει. Και εντάξει, ε, θα πρέπει λοιπόν από τη στιγμή που διαπραγματευόμαστε τότε προσφέρουμε, κάνουμε παραχωρήσεις. Αυτά λοιπόν και από το ΕΛΚ και το είπαμε και το είπε πολύ σωστά ο κ. Καπκαστάμκος, υποστηρίζουμε συγκεκριμένα τις ε, μακρινές ε, περιφέρειες ε, και το θέμα της μπανάνας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές τις εξαιρέσεις και να δούμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια όλοι κάτι θα πρέπει να παραχωρήσουμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περισσότερο πέρα από τις τροπολογίες μας και να προχωρήσουμε ώστε στο ε, να δούμε τι θα γίνει με τις εμπορικές συμφωνίες ε, που θα πρέπει να τις συντάσσουμε για αυτές τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές με ιδιαίτερη προσοχή και ταυτόχρονα ε, να, σε ορισμένου τομεί οι ζημίε που θα κάνουν και αναφέρομαι στην μπανάνα, πώ θα υπάρξει εκεί μια αντιστάθμιση. Λοιπόν, ε, εμεί νομίζω ότι με, πέρα, μαζί με αυτή την συμφωνία εμεί συντάξαμε μια ε, συμβαστική τροπολογία. Καλή είναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι εδώ όπω και αλλού ότι είναι συγκεκριμένη η συνθήκη τη Αβώνα σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτή την ειδική περίπτωση των εξόχων απομακρυσμένων περιοχών και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε όλοι ένα βηματάκι προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάτο που ήταν ιδιαίτερα σαφέ το μήνυμά σα και νομίζω και παράλληλα πήγαινε με αυτό που πήγε, έλεγε και ο κύριο Παπαστάμκο, ο εισηγητή. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει συζήτηση. Θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι θέσει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ έχουν αλλάξει και υπάρχουν πολλά νέα εισερχόμενα κράτη τα οποία έχουν επιρροή και κάνουν προτάσει που είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα λαμβάνονται υπόψη τα ε, ε, συμφέροντα τη Γεωργίας. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Γεωργίας να, να έχουν επιρροή. Εκπροσωπούμε την φωνή, είμαστε η φωνή του γεωργικού τομέα και γι' αυτό αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πιθανές συνέπειες στη Γεωργία πριν ε, πραγματοποιηθούν οι τελικές διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να μας αποκλείσουν πλήρως ε, επειδή έχουμε πολλά νέα κράτη που έχουν μεγάλη επιρροή. Αν θέλουμε να θέσουμε ε, εμπόδια, τελικά θα χάσουμε και θα χάσουμε την επιρροή μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις, να έχουμε λόγο, αλλά ταυτόχρονα να μην εμποδίσουμε τελείως τα πράγματα, μην τα μπλοκάρουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα πρότυπα και τις απαιτήσει μας, να μην είμαστε επίμονοι, υπερβολικά επίμονοι και να λέμε ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα θέλουμε εμείς. Γιατί τελικά θα αποτύχουμε μοιραία. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά για να δούμε πώς θα πετύχουμε τα ψηλότερα δυνατά πρότυπα αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουν και οι αγρότες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του αυτή και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους οι οποίοι και κατέθεσαν τροπολογίες αυτήν την έκθεση. Σημαντικό είναι, όπως το είπε και πολύ σωστά ο εισηγητής, να εξασφαλίζουμε τη συνοχή ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Ο γεωργικός τομέας, όπως υπόθηκε άλλωστε και αρκετές φορές εδώ στην Επιτροπή, δεν θα πρέπει να είναι ο χαμένος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Δεν μπορούμε να ζητάμε τα πάντα όλες τις παραχωρήσεις από τον γεωργικό τομέα. Σημαντικό είναι λοιπόν να πετύχουμε ένα δίκαιο ε, διεθνές εμπόριο δίκαιο και για τους ευρωπαίους παραγωγούς και για τους παραγωγούς βέβαια από τρίτες χώρες. Πολύ σημαντικό είναι οι διαπραγματεύσεις της, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ε, θα πρέπει να είναι σωστές αυτές οι διαπραγματεύσεις γιατί δεν μπορεί, θα πρέπει να υπάρξει μία υιοθέτηση ενός δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να προσέξουμε να μην επηρεάσουμε αρνητικά τις εμπορικές και οικονομικές δομές. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει και επιστημιστικό πρόβλημα μεγάλο και βέβαια από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες πρέπει να ανταποκρίνονται στα ίδια ποιοτικά προσόντα όπως τα κοινοτικά προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να παράχουν προϊόντα υψηλού κόστους και υψηλής ποιότητας, τα οποία συνεχεία θα υπονομεύονται από υποβασμισμένες εισαγωγές. Δεν επιτρέπεται εδώ να εφαρμόσουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ε, προϊόντα υψηλής ποιότητας θέλουμε να προσθέσουμε, να προσέξουμε τα πρότυπα και στην ευζοία στον ζώο, στην εκτροφή, στην παραγωγή, μέχρι και στην προστασία του καταναλωτή να εφαρμόζουμε προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις στο γύρο της Ντόχα να ολοκληρωθούν επιτέλους. Η κυρία Γέγκαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και το συνάδελφο κύριο Παπαστάμκο και σε όλους τους προλαλήσαντες. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα. Κατά την άποψή μου έχουμε δύο εταίρους να αντιμετωπίσουμε. Δεδομένου ότι εδώ μιλάμε κυρίως για διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Η Κομισιόν βασικά κάνει τις διαπραγματεύσεις και το Συμβούλιο, αλλά κυρίως η Κομισιόν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και εσωτερικά θέματα να λύσουμε, πώς θα προχωρήσουμε μέσα στο Κοινοβούλιο, ίντα, ε, αγροτική πολιτική. Εχθές ήμουνα στα ανθρώπινα δικαιώματα και άκουσα προβλήματα από εκεί και πώς θα μπορέσουμε εγκαίρως να φέρουμε τους συνομιλητές μας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Αυτό που ζω κάθε μέρα με την αντιπροσωπεία του Καναδά που δεν ε, εξελίσσονται ικανοποιητικά οι συζητήσεις, δεν με καθιστούν αισιόδοξοι στο τέλος θέλουμε και οι δύο πλευρές να κερδίσουν αλλά μας παρουσιάζουν τις αποφάσεις έτοιμες, ενώ θα έπρεπε και οι δύο πλευρές να κερδίζουν ισοδύναμες. Όσον αφορά τώρα τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, πρέπει να πούμε, ωραία, τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι σαυμάσια, άρα θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισοδυναμία αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας. Δεν μπορεί να έχω έναν τομέα εμπορίου ο οποίος προωθεί τις εξαγωγές και από την άλλη πλευρά θα πούμε «Α, στον αγροτικό τομέα ο επίτροπος, ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να ξοδέψει χρήματα για να καλύψει τα προβλήματα τα οποία υπονομεύουν τη θέση των Ευρωπαίων αγροτών». Εγώ πιστεύω ότι θα θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τις τροπολογίες για να επιφέρουμε ισοδυναμία. Ισοδυναμία. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε όλο και λιγότερο τους αγρότες μας, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως ας πούμε στην Αμερική, οι αγρότες υποστηρίζονται όλο και περισσότερα. Άρα θα πρέπει λοιπόν να ξεκινάμε τη συζήτηση των θεμάτων με τους συνομιλητές μας νωρίς. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που οι τροπολογίες έφτασαν σε εμά νωρίς, εγκαίρως. Ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρέπει εκ των προτέρων να καθορίσουμε τη θέση μας για να είμαστε έτοιμοι διότι το, το Κοινοβούλιο ή θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει, θα απορρίψει την εμπορική συμφωνία. Το ίδιο ισχύει για την Κορέα, για το Μαρόκο, για το Μερκοσούρ, που θα μας επηρεάσει πολύ σημαντικά και για τον Καναδά. Εντάξει θα μου πείτε κάθε διμερή συμφωνία δεν είναι και τόσο όγκο, αλλά άμα τι πάρουμε όλες μαζί θα δείτε ότι οι επιπτώσεις είναι σημαντικότατες. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε και πιστεύω ότι με τις τροπολογίες έχουμε μια θαυμάσια έκθεση στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ισαμπέδ. Πόλσεν, Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπαστάμκο συνέταξε μια, ένα καλό ξεκίνημα για κάτι που τελικά θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι το θέμα γίνεται πολύ σοβαρό. Όλο και περισσότερες διμερείς συμφωνίες συνάπτουμε πλέον. Αυτό είπε και η κυρία Γέγκλα. Σε κάθε σημείο χωριστά δεν μοιάζει το θέμα να είναι επικίνδυνο. Πρέπει όμως να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συνολική συμφωνία που όλοι να μπορέσουμε να τηρήσουμε. Αρχικά, ίσως τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο δύσκολα από το να είχαμε μία μόνο συμφωνία με, τη Μερκοσ... με τις χώρες Μερκοσούρ. Όμως, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θεωρώ ότι όλο και περισσότερα χάνουμε, όλο και περισσότερα παραχωρούμε. Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ κάτι πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι γενναιόδορη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη στον χώρο της γεωργίας, ας πούμε στην Αφρική. Η Αφρικανική Ήπειρος πλέον κινείται εντελώς προς την λάθος κατεύθυνση και εμείς ο πλησιέστερος και πλουσιότερος τον τους δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να συνεχίσουν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο με το να χτίσουμε μια πολιτική γεωργίας η οποία να στηρίζεται ή να δυναμώνει από τη γενεοδορία μας. Τώρα, όταν δούμε όλες αυτές τις συμφωνίες, είτε περνούν μέσω του ΠΟΕ, είτε είναι διμερείς, υπάρχει κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. είναι το θέμα της φροντίδας που πρέπει να μας απασχολεί. Γι' αυτό, σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα στα θέματα, ας πούμε, της προστασίας της ευζοίας των ζώων. Πρέπει να έχει υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική αυτή τη πολιτική. Δεν είναι τι αισθανόμαστε μόνο και τι ε, σκεφτόμαστε όσον αφορά την ηθική, τη διοντολογία κλπ. Πρέπει να υπάρξει μια επιστημονική βάση στην πολιτική μας και μόνον έχοντας αυτή την επιστημονική βάση θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πραγματική πολιτική προστασία των ζώων που να είναι λειτουργική διεθνώς. Γιατί τελικά δεν ακούγεται πολύ πιστικό όταν συνεχίζουμε να μιλάμε μόνο για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλάμε μόνο για μα. λέμε «Α, κοιτάξτε εμεί πώ αγαπάμε τα ζώα μα, του τους τι αγελάδε κλπ». Αλλά είναι αυτά θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη παγκοσμίω τα θέματα της υγείας των ζώων και της ευζοίας των ζώων πρέπει να συνδεθούν ξεκάθαρα με πολιτικές υγείας, με το δικό μας μέλλον, με τρόπο πολύ πιο δυνατό από ό,τι συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια διεθνή συμφωνία αφενός, πρέπει αφετέρου να δουλέψουμε δείχνοντας αλληλεγγύη στους στοχότερους λαούς του κόσμου και τρίτον πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς κοινή νομοθεσία η οποία θα είναι μια νομοθεσία που εμεί θα μπορούμε να στηρίξουμε με κάθε σοβαρότητα στις ε, διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Γιάρ. Και μετά η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Παπαστάμκο για αυτή την έκθεση την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική. Πιστεύω ότι η έκθεση και οι τροπολογίες βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μερικές εισαγωγικέ παρατήρησεις. Βεβαίω, η καλύτερη συμφωνία θα ήταν μια διεθνή ε, Διμερείς, πολυμερεί συμφωνίε είναι πάντοτε δεύτερη σε σειρά προτεραιότητο. Πιστεύω δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες να επιτύχουμε μια παγκόσμια διεθνή συμφωνία. Πιστεύω ότι οι καλύτερες ε, εμπορικές συμφωνίες είναι εκείνες οι οποίες δεν δημιουργούν, ε, δεν καθιστούν αποζημιώσεις υποχρεωτικές. Και θα μπορούσα επίσης να πω ότι με τις συμφωνίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα η μία πλευρά παίρνει μία θοδέσμη η άλλη μία πλευρά παίρνει αποζημίωση. Ε, αυτές οι αποζημιώσεις, το compensation, ε, δημιουργούν συνέχεια προβλήματα ε, διότι αναγράφονται και στον τύπο, έχουν οικονομικές επιπτώσεις και πιστεύω θα ήταν καλύτερο εάν κλείσουμε συμφωνίες που, όπου δεν αναφέρονται καθόλου οι αποζημιώσεις. Δεύτερον, εάν διαπιστώνουμε ότι έχουμε κλείσει συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν μειονεκτήματα, βάζουν σε μειονεκτική θέση τους παραγωγούς μας, τότε βέβαια πρέπει να τους αποζημιώσουμε. Όταν διαπιστώνουμε, όταν έχουμε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις στα ίδια πρότυπα Πρέπει όμως και εμείς να προσέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διατυπώνουμε και επιβάλλουμε καινούργια πρότυπα, καινούργιες προδιαγραφές, αν αυτές μπορούν να λειτουργήσουν στο διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές δημιουργούνται αντιφάσεις. Ε, δεν ασχολούμαστε μόνο με τη δική μας ευημερία. Λειτουργούμε σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει πάντοτε να κοιτάμε τι πρότυπα και τι προδιαγραφές ισχύουν στα άλλα μέρη του κόσμου, εκτός από εμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαγκίνες τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον εισηγητή, τον κύριο Παπαστάμκο για την έκθεση αυτή. Ε, έχω μια συγκεκριμένη τροπολογία που ελπίζω να λάβετε υπόψη που αφορά τις μελέτες επιπτώσεων και αντί να κάνουμε μια συνολική και ξεπερασμένη έκθεση από πλευράς κομισιών, Θέλουμε μια ε, έκθεση συγκεκριμένη για τον τομέα και που να, μελετάει τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένο υποτομέα, ας πούμε το τομέα του βοήου κρέατος. Τώρα, στο θέμα των αποζημιώσεων, διαπιστώνω ότι αυτοί που αποζημιώθηκαν για την μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης προτιμούν να καλλιεργούν σαχαρότευτλα ακόμα. Το θέμα της αποζημίωσης είναι ένα χρυσωμένο χάπι που μετά σου αφήνει μια εξαιρετικά πικρή γεύση γιατί δεν έχει τίποτα να κάνεις στην εκμετάλλευσή σου. χάνει μια ολόκληρη επιχείρηση και κάποιες χώρες χάνουν έναν ολόκληρο κλάδο. Ας είμαστε απολύτως σαφές, σαφείς. Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού ε, ε, για το επόμενο έτος εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας. Που πού προέρχονται οι, δια, οι αποζημιώσεις όταν επιβάλλονται τόσο σοβαρές περικοπές στον προπολογισμό μας. Τρίτο θέμα. Υπάρχει μια πολιτική επιταγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σοβαρή με το θέμα της ε, διατροφικής ασφάλειας. Ιδάλλως πρέπει να εγκαταλείψουμε τη γεωργία. Υπάρχει μια πορεία στον τομέα αυτό, όχι που να με ικανοποιεί πάντα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε. Όταν αρχίζουμε να στηριζόμαστε στους παραγωγούς τροφίμων, τροφίμων από τις τρίτες χώρες θα σταματήσουμε, μπορεί να σταματήσουν οι εξαγωγές και τότε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Επανέρχομαι στο θέμα της αγοράς αχάρεως αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις, την ποιότητα ε, της ζάχαρης που απαιτούμε στις ποσότητες που θέλουμε και έχουμε πρόβλημα για του χρόνου. Άρα υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων που αφορούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελευταίο, θέλω κάτι να ταράξω λίγο τα νερά εδώ, γιατί γίνονται προπολογισμοί, ψηφοφορίες κτλ. Μιλάμε για τα πρότυπα ευζοία των ζώων και ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Πόλσον όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, ενδιαφέρονται ε, τόσο πολύ ε, για αυτό το θέμα της ευζοής των ζώων όσο λέμε εμείς μερικές φορές. Ακούμε πολλές φορές, ακούω εγώ πολλές φορές το πολύ ε, θορυβόδες λόμπι της προστασίας των ζώων ενώ άλλοι που παλεύουν για το εισόδημά τους μου λένε άλλα ως, ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θορυβούν αλλά εμείς σε αυτή την Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια χρόνια κατάσταση για τους παραγωγούς αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν ένας από αυτούς που ψήφισαν για το θέμα των κλοβών ε, στην, ε, ε, στην ε, νομοθεσία για τα ζώα θα το καταψήφιζα τώρα και ας με καταδικάσουν. Το σύστημα λειτουργεί γιατί παράγονται αυγά καλής ποιότητος σε καλή τιμή. Τώρα ε, ε, ξοδεύουμε δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθούμε σε νομοθεσία ευζοίας των ζώων που για την οποία δεν υπάρχει ημερομηνία στόχος. Δηλαδή επιβάλλουμε τεράστιο κόστος. Το ξέρουν οι Γερμανοί τι συνέβη στη χώρα τους είναι οι καλοί άνθρωποι της Ευρώπης και εισήγαγαν τα πρότυπα αυτά εκ των προτέρων και τώρα πέφτει η παραγωγή τους και εισάγουν αυγά από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπόλοιπη Ευρώπη ή από άλλες περιοχές αυγά Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή αυτά τα ζητήματα θα ε, ε, βαθύνουμε την κρίση. Δεν ακούω διαμαρτυρίες από τους, πολίτες για τα θέματα της ε, ευζώειας. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο ζώα, αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί Εξάγουμε την ε, παραγωγή ε, ε, εξάγουμε τρόφιμα επειδή τα, έχουμε πνίξει στους περιορισμούς. Αυτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο για αυτή την έκθεση, γιατί ξέρω ότι είναι σε καλά χέρια η έκθεση αυτή. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, απλώς να τονίσω ότι υποστηρίζω όλους ότι ο υπολογισμός, η εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και έγκαιρα. Βεβαίως καλύτερα θα ήταν να συνεχιστεί ο γύρος της Ντόχα και μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Ε, προ, προτιμώ την Τόχα και τον ΠΟΕ από τις διμερείς διαπραγματεύσεις διότι συνήθως στις διμερείς συμφωνίες πολλές φορές εμείς είμαστε οι χαμένοι. Τώρα όμως διαφωνώ με την παρατήρηση που έγινε ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο γενναιόδοροι με την Αφρική. Ε, ε, Βεβαίω ο τύπος αναφέρει συνέχεια προβλήματα αυτής της Υπήρου, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήδη το 90% των εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων της Αφρικής έρχεται σε εμά. Ήδη είμαστε λοιπόν πάρα πολύ γενναιόδοροι. Είμαστε η αγροτική Ήπειρος ε, ε, στο, στο, στην Ιφίλιο που δείχνει τη μεγαλύτερη γενοδορία έναντι της Αφρικής. Όσον αφορά δε την ε, ευζοία, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το δημιουργήσαμε ήδη και πιστεύω ότι ότι έχουμε ένα περιθώριο συζήτηση σε αυτό το θέμα. Εκεί που δεν θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμού καθόλου είναι στην ασφάλεια των τροφίμων. Ε, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Οι διαπραγματεύσει μα εδώ πρέπει να είναι πολύ σκληρέ. Δεν είναι λογικό στην Ευρώπη να απαγορεύουμε ε, ε, φυτικά προϊόντα ε, για την προστασία των καταναλωτών ενώ ανοίγουμε παραθυράκια εισαγωγών ε, διότι εισάγονται προϊόντα από χώρες όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα ε, φυτοφάρμακα ή προϊόντα τα οποία δεν εγκρίνουμε εμείς πρέπει οπωσδήποτε να επιβάλλουμε ένα ποιοτικό έλεγχο εισόδου ε, εφόσον έχουμε ποιοτικό έλεγχο εξόδου, δηλαδή εξαγωγών, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία στο ποιοτικό έλεγχο εισαγωγών. Ναι, να πουλάνε τα προϊόντα τους στην Ευρώπη, αλλά να έχουμε ίδιες προδιαγραφές, ίδια πρότυπα, χωρίς να υπονομεύουμε τη δική μας παραγωγή. Και επανέρχομαι στο θέμα της ε, προστασίας των ζώων. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές έχω λιγότερη εμπιστοσύνη σε ορισμένες εταιρείες προστασίας ζώων. Επί 20 χρόνια ακούω την, το ίδιο Ευαγγέλιο, οι μεταφορές των ζώων, πώς θα γίνονται, δεν γίνονται σωστά, είναι χάλια, υποφέρουν κλπ. κλπ. Τώρα ε, έρχονται ε, ζώα σε εμά τα οποία έχουν μεταφερθεί από περιοχή περιοχή της Βραζιλίας, της Αυστραλίας όπου δεν μπορούμε να ελέγξουμε ε, πώς ακριβώς μεταφέρονται και με ποιες συνθήκες μεταφέρονται τα ζώα σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση και να μάθουμε από τα παθήματά μας. Τα μαθήματά μας να μας γίνουν πάθημα. αυτή η όλη ιστορία της προστασίας των ζώων και των τόσο αυστηρών ε, προδιαγραφών λόγω της πίεσης ε, όλων αυτών των συλλόγων ε, και προστασίας των ζώων έχει δημιουργήσει μια αρνητική κατάσταση ενώ εμείς προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε στα συμφέροντα των Ευρωπαίων αγροτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντες. Ο κύριος Νίκολσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ο τομέας αυτός που συζητάμε σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικός και πραγματικά ε, με ευχαρίστησε πολύ αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαστάμκο για την εξαιρετική του έκθεση η οποία μας ε, στρέφει προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει νομίζω όλοι να παραδεχτούμε ότι μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία του ΠΟΕ οι διμερείς συζητήσεις θα συνεχίζονται. Και το αν και κατά πόσον ε, είναι καλύτερη η μια συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ που να μπορούμε όλοι την προσυπογράψουμε ή αν θα συνεχίσουμε να έχουμε ξεχωριστές ε, απόψεις και συμφωνίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες περιοχές, αυτό είναι κάτι που όλο και περισσότερο θα τεθεί υπό συζήτηση. Γιατί ποιο μπορεί να είναι, ε, μπορεί να υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα αν είναι θετικές διαπραγματεύσεις, αλλά θετικές για ποιον. Κατά την άποψή μου, οι διαπραγματεύσεις πάντοτε ε, καταλήγουν θετικά στον τομέα της γεωργίας. Οι αγρότες σε κάθε περίπτωση έχουν θυσιαστεί από τους διαπραγματευτές και αυτό είναι ένας από τους σοβαρότερους φόβους μου και πιστεύω ότι και πολλοί άλλοι θα συμφωνούν μαζί μου ότι πάντοτε οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα για το όφελος των συζητήσεων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη συζήτηση για, την, ε, για το βοδινό από την Βραζιλία και τη συμφωνία σε επίπεδο Μερκοσούρ και τι μπορεί να υποφεληθούμε. Τα πράγματα φυσικά έχουν εξελιχθεί και ε, εξ όσων αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή η τιμή του βοηού κρέατος στη Βραζιλία είναι η ίση με αυτή που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά έκτοτε, τα πάντα ρί, τίποτα δεν μένει ίδιο παρά τις δυσκολίες που έχουμε. Υπάρχουν τομείς ε, τους οποίους έχω πολύ συγκεκριμένες πεπιθήσεις. Ας πούμε τα πρότυπα που εφαρμόζουμε εδώ είτε πρόκειται για εισαγόμενα είτε για εξαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι τα ίδια, τα ίδια πρότυπα. Ένα αυτοκίνητο που δεν ε, ανταποκρίνεται στα πρότυπά μας δεν μπορεί να μπει. Γιατί να μπαίνει η τροφή λοιπόν χωρίς να ανταποκρίνεται στα πρότυπα και πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ε, ε, ε, σε αυτούς με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή ότι αν περάσουν αυτό το όριο εμείς θα είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξεκάθαρα. Δεν θα το κάνετε εάν δεν τηρήσετε αυτό τον κανόνα. Η Μέρουντ Μαγκίνες εισήγαγε στη συζήτηση ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όλοι να ακούσουμε. Έχει δίκιο. Ε, και αυτό μπορείς να το πας και πιο πέρα από το θέμα της ευζοίας των ζώων, να μιλήσουμε και για την ε, το περιβάλλον. Μίλησες για πράσινη γραφειοκρατία. Μιλάμε όλοι για κόκκινη γραφειοκρατία, red tape, αλλά υπάρχει και η πράσινη γραφειοκρατία. Η ΚΑΠ ε, προχωρεί επειδή κάποιοι 5.000 ε, άτομα ζήτησαν να γίνει πιο πράσινη, ε, πράσινος ένας πυλώνας. Δηλαδή 5.000 άτομα μας ζητάνε κάτι και εμείς κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν. πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει Μέιρετ. Είναι τόσοι άνθρωποι που δεν, μπορούμε, δεν μπορούν καν να αγοράσουν το φαγητό που παράγεται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν διαδικασίες που έχουν επιβληθεί συν το χρόνο και τις έχουμε ψηφίσει εμείς και πρέπει τώρα να τις εφαρμόσουμε και θα προκληθεί αυτό που λέμε ότι το 2012 θα υπάρχουν 83 εκατομμύρια αυγά την ημέρα τα οποία θα καταστρέφονται. Εν τω μεταξύ άλλοι άνθρωποι πεινάνε. Τι θα γίνει με αυτά τα αυγά. Υπάρχει ένα δίλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει αντιμετωπίσουμε τώρα και θα έρθει η Κομισιόν και θα μας πει «Α, δεν είσαι καλό παιδί, θα σου βρούμε 5.000 ευρώ». Α, τι λες, δεν αρκεί, δεν αρκεί. Διότι ακούσαμε από άλλους συναδέλφους στη Γερμανία και τις κατοχώρες και αλλού που έχουν εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία. Δεν μπορεί τώρα να τους ζητήσουμε να πληρώσουν τίμημα επειδή ήταν καλά παιδιά ε, ε, έγιναν αυτά τα οποία του, έκαναν αυτά τα οποία του ζητήθηκαν πριν το επόλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είμαστε σε νέα πραγματικότητα, χρειαζόμαστε νέα πραγματικότητα για να προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω επ' αυτού πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο μέλλον. Ευχαριστώ, Κεν Νίκολσον. Η κυρία Πατρονέβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω όλα αυτά που υπόθηκαν γι' αυτό, ότι απαιτούνται συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών μας απέναντι στους παραγωγούς άλλων χωρών αναφέρθηκε η προστασία του περιβάλλοντος, η ευμάρεια των ζώων, όλα αυτά. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και τη δημιουργία προδιαγραφών, την οθέτηση προδιαγραφών για την γεωργική ευρωπαϊκή παραγωγή. Μέτρα που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι υπόλοιποι δεν σέβονται και μπορούν έτσι να εξάγουν ελεύθερα σε εμά τα προϊόντα τους χωρίς αυτούς τους περιορισμούς και θα ήθελα να πω ότι έχουν δίκιο όλοι όσοι είπαν πριν από μένα όλα αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε έτσι να έχουμε ε, κάτι ε, που να βαρύνει από την άλλη μεριά απέναντι σε κάθε εμπορική συναλλαγή, σε κάθε εμπορική συμφωνία. Ε, δεν θα πρέπει να θίγουμε έτσι, να ζημιώνουμε την ε, γεωργία μας. Ο πλέον στην υπόθηκε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν ιδιαίτερα αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και ακριβώς η γεωργία τους καλύπτει μια περιορισμένη έκταση και υπάρχει και ένα πρόβλημα διαφοροποίησης. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να αλλάξουν σε λογικά τουλάχιστον χρονικά πλαίσια την καλλιεργιά τους. Άρα λοιπόν ε, γι' αυτό και έχουμε κλείσει ιδιαίτερες συμφωνίες με εκείνους. Ε, τώρα, πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν εδώ, θα ήθελα να πω, να προσθέσω και κάτι ακόμα, μία ακόμα πτυχή στην όλη μας συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Παπαμστάμκο να τα συλλογιστεί αυτά, τα σκεφτεί αυτά. Βέβαια, θα ήθελα ταυτόχρονα να του δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Παπαστάμκο για τον ιδιαίτερα θετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα ζωτική σημασία για όλου εμά σχετικά με όλα τα προβλήματα της γεωργίας. Θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο γίνεται ευρύτερα, ένα ευρύ ορίζοντα και ιδιαίτερα καλά διαρθρωμένα. Δεν μπορούμε έτσι εδώ και εκεί αποσπασματικά να αφιερούμε την προσοχή μας εδώ και εκεί επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να έχουμε μια γενική σφαιρική εικόνα του όλου θέματος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο των προβλημάτων της γεωργίας όπως επίσης και της τροφικής αλυσίδας από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Έτσι. Θα πρέπει να, αν να μιλήσουμε σοβαρά για την κυρία πολιτική μέχρι το 2020 και αν θέλουμε να δούμε ταυτόχρονα τι λέει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Να μην μιλάει μόνο για εμπορικά μέτρα και διεθνές εμπόριο αυτή η ανακοίνωση. Οι προθέσεις είναι καλές, παρά τις καλές προθέσεις, παρά τις προτάσεις που υποβάλλονται. Εάν συνεχίσουμε εμείς να αναθεωρούμε την κοινή γεωργική πολιτική και να επηρεάζουμε μόνο από τη μια μεριά, από τη μια άκρη τα πράγματα, τότε θα αποτύχουμε δεν θα διαθέτουμε μια γεωργία με πραγματική δυνατότητα αηφόρου ανάπτυξης μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε επίπεδο αγοράς και διεθνούς εμπορίου θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν υπάρχουν προοπτικές όμως για αυτά στα πλαίσια της ΚΑΠ για το 2020. Η έκθεση την οποία τώρα συζητάμε αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάνιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες και τον κύριο Νίκολσον. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι όταν έχει μια συμφωνία με ένα άλλο εμπορικό μπλοκ, ε, είναι η, εφαρμογή, η υλοποίηση ναι, τους λέμε ότι ναι βεβαίως ε, ε, ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε τα δικά σας πρότυπα, μας λένε οι, οι τρίτοι δηλαδή εταίροι και ελάτε εδώ στην Αργεντινή να σας δείξουμε τι ωραία που εκτρέφουμε τα ζώα μας κλπ. Ε, πάμε λοιπόν εμείς μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, μας πάνε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μας ποτίζουν, μας ταΐζουν καταπληκτικά, μετά βλέπουμε και ένα ωραίο σοου και μας δείχνουν και το αγρόκτημα και όλα είναι θαυμάσια. Εν τω μεταξύ η κανονική δουλειά γίνεται 400 χιλιόμετρα μακριά από την πρότυπη μονάδα όπου τα ζώα όπου τα ζώα βρίσκονται σε κακές συνθήκες και όπου βεβαίως οι προδιαγραφές δεν ε, τηρούνται. Δεν μπορεί να πει κανείς κοιτώντας ένα βούτυρο, ένα πακέτο βούτυρο ότι το ζώο που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν το έχουμε δει ποτέ ότι έχει τύχη καλής μεταχείρισης. Βεβαίως θέλουμε τα πρότυπα αυτά εγώ είμαι πάντοτε σε ένα δίλημα όταν κάνω αυτές τις επισκέψεις. Λέω να πάω πιο μέσα στη χώρα και να δω τι γίνεται πραγματικά στις μονάδες εκτροφών. Αλλά δεν, μας, ούτε, δεν έχουμε τον καιρό και δεν θα μας αφήσουν κιόλα. Δεν θέλω να δούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάτι μου λείπει γιατί δεν μπόρεσα εγώ να απολαύσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που μόλι είπε προηγουμένως ο μιλητής. Αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Ε, το είδα, το, το είδα, το διάβασα, το άκουσα όπως πρέπει. Θα θα χαιρετήσω την εργασία του συναντέλφου κύριου Παπαστάμκο. Η εργασία του, η συνεργασία με συνεργά όλων μα με τι απόψει όλων μα, με τι θέσει που εκφράσαμε όλοι μα με τι τροπολογίε ε, που προτείνεται να ληφθούν υπόψη, νομίζω ότι δείχνουν ακριβώ μια ανάκληση τη άποψη ε, εδώ και 18 μήνε τη επιτροπή μα σε αυτό το θέμα. Και πριν να πάμε στην Αργεντινή και στην Βραζιλία, πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα στο σπίτι μα να δούμε πώ συνάδελφοι όλοι θα κατανοήσουν ότι αυτό το άνοιγμα και η ανάπτυξη και σε άλλους οικονομικούς τομείς μπορεί να επιτευχθεί μόνο εις δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος ενός τομέα που έχει μεγάλη σημασία για διατροφή των Ευρωπαίων γιατί εντάξει εξάγουμε αλλά πρώτα απ' όλα παράγουμε για τον εαυτό μας και αν μέσω των εισαγωγών εμείς ε, σκοτώνουμε, φωνεύουμε τους παραγωγούς μας δεν διακινεται μόνο η θέση μας στην διεθνή αγορά αλλά και η ανεξαρτησία της της διατροφής στην Ευρώπη, η τροφική αλυσίδα η οποία κινδυνεύει. Και θυμάμαι ο αρμόδιος επιτεμπορίου Επίτροπο το τι είχε πει στο Μεκέκλειο, δεν θυμάμαι που το είχε πει αυτό στο Βρυξέλλε ή στο Στρασβούργο. Έλεγε ότι αυτέ οι διαμαρτυρίε μα δεν είχαν κανένα νόημα. Έτσι κι αλλιώ κάπου θα, από κάπου θα το αντισταθμίζαμε εδώ στην Επιτροπή. Ε, είναι σημαντικό και να υπενθυμίσουμε κ. Ντεγκούχτο, δεν γίνεται έτσι εύκολα αυτή η αντιστάθμιση. Βέβαια, μπορούμε κάποιον να αποζημιώσουμε από τη στιγμή που θα υποστεί λίγη ζήμια, αλλά όταν ε, θέλουμε να αντικαταστήσουμε μια παραγωγή απλά και έτσι μόνιμα. Και όταν έχει καταστραφεί πάνω από το 5% η παραγωγή, δεν έχουμε δυνατότητα οικονομική σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντισταθμίσουμε, να αποζημιώσουμε τους ε, ε, παραγωγούς. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι μέλη εδώ στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ακριβώ και η Επιτροπή και νομίζω ότι ε, ο επίτροπο για τη Γεωργία μπορεί, θα μα υποστηρίξει σίγουρα το σύνολο τη Επιτροπή επιτέλου να καταλάβουν ότι αν προχωράμε από τη μία θυσία στην άλλη τι θα γίνει και η θέση μα στις παγκόσμιε αγορέ θα περιοριστούν αυτέ τι θέσει, αλλά και η ίδια η Γεωργία ε, η Ευρωπαϊκή θα θυσιαστεί. Ευχαριστώ, κύριε Ντόντα. Ο κύριος Ντανέλη. είναι ο τελευταίος ομιλητής που έχω στον κατάλογο των αγορητών και μετά θα περάσουμε στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Γιώργο και όσους ασχολήθηκαν με εξαιρετικό τρόπο ε, για ένα ιδιαίτερος ε, κρίσιμο αλλά και δύσκολο θέμα. Ε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ε, και κοινά αποδεκτό και βεβαίως ε, ένα παραπάνω από την αριστερά ότι θα πρέπει να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη και να στηρίζουμε με κάθε ε, εύλογο τρόπο τους λαούς των τρίτων χωρών και κυρίως βεβαίως τους χυμαζόμενους της Αφρικής. Φοβάμαι όμως ότι στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών μας ή του ΠΟΕ κάνουμε σημαντικές εκπτώσεις στο όνομα αυτής της αλληλεγγύης αλλά για ιδιωτελείς και κοινικούς και υποκριτικούς λόγους ε, κάνουμε ιδιαίτερες εκτόσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφική ασφάλεια των προϊόντων, των διατροφικών αλλά και με, την μη αηφόρο διαδικασία ε, παραγωγής τους. Αυτό είναι και σε βάρος του καταναλωτή βεβαίως αλλά Επίσης ε, νομίζω ότι εάν ε, δεν έχουμε υπόψη μας ότι με αυτόν τον τρόπο ε, δημιουργούμε συνθήκες αθέμητου και ανήθικου ανταγωνισμού στους Ευρωπαίους παραγωγούς οι οποίοι παραπέουν συνεχώς νομίζω ότι χάνουμε ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ενδιαφερθούμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε. Ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή σήμερα έχει το λόγο. το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω τις εντυπωσιακέ τροπολογίες, ε, το αριθμό τροπολογιών που έχουν προταθεί δίνει, δείχνει και τη σημασία της έκθεσης ε, για την Επιτροπή αλλά και τη σημασία του θέματος. Θέλω να σας ενημερώσω τις πρόσφατες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Με βάση τα τελευταία δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπολογίζουμε ότι το 2010 οι εξαγωγές μας φτάνουν σε ιστορικό ρεκόρ αναμένουμε ότι θα ξεπεράσουν τα, ε, τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δύο τρίτα αυτών των εξαγωγών θα είναι ε, τελειωμένα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και επεξεργασμένα προϊόντα. Μόνο το 8,5% θα είναι πρώτε ύλε, δηλαδή ε, γεωργικά προϊόντα. Επίση, περιμένουμε ότι το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο θα είναι θετικό επιβεβαιωθεί αυτό. Θα είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Η προηγούμενη ήταν το 2006 που είχαμε και πάλι θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Αυτό θα επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη τάση βελτίωσης του εμπορικού μας ισοζυγίου. Έτσι λοιπόν τα πράγματα φαίνεται ότι μπαίνουν και πάλι σε καλό δρόμο μετά από την ε, μεγάλη αύξηση ε, και την πτώση των ε, γεωργικών τιμών που έγινε την περίοδο από το 2007 έως το 2009. Επίσης, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2010 αναμένεται να είναι υψηλότερες από ότι οι συνολικές γεωργικές εξαγωγές για κάθε έτος προ του 2002. Αυτή η κατηγορία μοιάζει ότι είναι το πιο ε, δυναμικό κομμάτι των εξαγωγών μας. Και τώρα έρχομαι στο σχέδιο έκθεσης και στις τροπολογίες θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω τις σκέψεις μου με ε, και να τις χωρίσω σε κάποιες κατηγορίες. Πρώτο θέμα αφορά την σωστή ισορροπία όταν συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες στο χώρο της γεωργίας και μεταξύ γεωργίας και άλλων τομέων. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι θεώρησαν ε, κατάλληλο να αντικαταστήσουν τον, όρο condemns με κάτι άλλο. Παράγραφος 3. Επίσης η, η Κομισιόν διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες ε, με τη βάση διαπραγματευτικών οδηγιών οι συνήθως θέτουν στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί ισορρόπες και ολοκληρωμένες συμφωνίες με τους εταίρους μας με στόχο την απελευθέρωση, ουσιαστική απελευθέρωση όλου του εμπορίου. Δεύτερο θέμα αφορά την εφαρμογή των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εισαγόμενα αγαθά. Θέλω να υπογραμμίσω και για μία ακόμα φορά ότι τα ε, προϊόντα ε, από αγροτικά τρόφιμα που ε, περιλαμβάνονται εδώ πρέπει να συμμορφώνονται με τη ε, ε, νομοθεσία εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των φυτών και των ζώων. Ενώ πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές συνάδουν με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας δεν μπορούμε ε, να επιβάλλουμε σε τρίτες χώρες διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής όπως παραδείγματος χάρη πρότυπα στην ευζοία των ζώων στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στα πλαίσια του ποε. η ευρωπαϊκή ένωση συνεχίζει να πιέζει για καλύτερη αναγνώριση αυτών των προτύπων στα κατάλληλα διεθνή φόρα. επίσης επιτρέψτε μου να κάνω μια πιο συγκεκριμένη παρατήρηση σχετικά. η συμφωνία μια SPS τι απαιτεί αντίστοιχα υγειονομικά ή φυτοϊγειονομικά ε, μέσα και όχι τα same, τα ίδια όπως προτείνονται σε κάποιες διαπραγματεύσεις και όπως επεσήμανε εξάλλου το ίδιο θέμα και ο εισηγητής μας. Τώρα, όσον αφορά το πολυμερές ε, σύστημα εμπορίας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ισχύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, με τους νόμους του 2002 και του 2008 ξεκίνησε προς την κατεύθυνση της στήριξης ε, στρέβλωσης του εμπορίου εξίσου ισχύει ότι στη, λόγω των υψηλών παγκοσμίων τιμών η, ε, ε, τα αποτελέσματα ήταν μικρά, κάτω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Τώρα όσον αφορά το τρίτο σκέλος του σχεδίου έκθεσης για τις πολυμερείς και διμερείς εμπορικές σχέσεις, θέλω να πω τα εξής. Πρώτον, σε σχέση με το, ε, την νομοθεσία του Καναδά για τον καπνό. Η Κομισιόν έχει θέσει το θέμα του νόμου C32 μαζί με άλλα μέλη του ΠΟΕ σε συνεδριάσεις του ΠΟΕ και πιο πρόσφατα στις συνεδριάσεις της 3ης και 4ης Νοεμβρίου φέτος. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στο θέμα αυτό η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά στις ανησυχίε που διατυπώθηκαν μέσω τροπολογιών για την έλλειψη ενημέρωση από πλευρά Κομισιόν για τι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσει, όπω α πούμε τον Καναδά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή ΙΝΤΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνεται τακτικά για τι τρέχουσε διαπραγματεύσει συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τον Καναδά. Θέλω επίση να υπογραμμίσω ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τα θέματα των δασμών με τον Καναδά το τρίτο σημείο που ετέθη ε, στη διάρκεια της συζήτησης αφορά τις αφρικανικές χώρες. Θέλω να επαναλάβω ότι με τις χώρες ΑΚΕ έχουμε ανοιχτά σύνορα. Έχουμε μια πολιτική χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις, χωρίς οποιοδήποτε δασμολογικούς περιορισμούς με τις χώρες ΑΚΕ. Επίσης, στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισής μας και στις συζητήσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ, η πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας. Επίσης, θέλω να επαναλάβω, όπως και υπογραμμίζεται και στην έκθεση, και όπως υπογράμμισαν και κάποιοι από τους ομιλητές, ότι οι επιδοτήσεις εξαγωγών ουσιαστικά βρίσκονται σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο αλλά ε, επαναλαμβάνουμε στους εταίρους μας του ποε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τις καταργήσουμε τελείως αυτές τις επιδοτήσεις εξαγωγών αν και εκείνοι είναι διατεθειμένοι να εξαλείψουν παρόμοια μέτρα που έχουν θεσπίσει όπως την επιστηστική βοήθεια ή ε, τις ε, εμπορικές κρατικές επιχειρήσεις. Τέλος, θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι σε πολλές τροπολογίες η ανάγκη ε, ε, συμμόρφωσης με τα συμβατικά μέτρα του ΠΟΕ υπογραμμίζεται και επίσης ότι είμαστε διατεθειμένοι και διαθέσιμοι να έρθουμε να συζητήσουμε μαζί σας οποιοδήποτε θέμα αφορά τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε το Διευθυντή κύριο και να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Παπαστάμκο για να, κατα... να πει τα τελικά. Κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει περάσει η ώρα. Θα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις... και βεβαίω να παραλάβω για τις ε, σημαντικές τροπολογίες τους. Ε, ξεκινώ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον αγαπητό κύριε Σιβένα και θέλω να πω ότι το καταδικάζω είναι μια γλώσσα πάρα πολύ λέξη αποδεκτή και στη διεθνή διπλωματία αλλά και στην ευρωπαϊκή διπλωματία και γιατί όχι δεν πρέπει να αφορά και την διαθεσμική λειτουργία και τη διαθεσμική σχέση. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς περνούν οι επίτροποι και εκπρόσωποι της Κομισιόν όταν επισκέπτονται την Αργεντινή ή την Βραζιλία ή άλλες χώρες, αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος ε, Άγνιου ή πώς συμπεριφέρονται οι διπλωματικές αποστολές, τα γραφεία δηλαδή αντιπροσωπείες της Κομισιόν σε τρίτες χώρες για τις οποίες ο Ευρωπαίος φορολογούμενος καταβάλει ένα σημαντικό ποσό και ο, ο ευρωπαϊκός ε, για αυτές τις αποστολές και πώς αυτές οι αποστολές διασυνδέονται ή όχι με τις κατατόπους κυβερνήσεις και αν εκπροσωπούν εκεί το ευρωπαϊκό συμφέρον ή άλλες καταστάσεις. Βεβαίως μας ενημερώνει, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που συμφωνείτε μαζί μου με το νεύμα σας. Και τι θα πει ενημερώνει η Κομισιόν την ίντα ή στέλνει περιορισμένα έγγραφα. Χάρη κάνει η Κομισιόν στην ίντα ή αύριο ενημερώσει την Επιτροπή ε, Γεωργίας του Κοινοβουλίου. Το ζητούμενο είναι αν λαμβάνει υπόψη τη θέσεις είτε τη ίντα είτε της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή τι είναι ο μεγάλος αδελφός, είναι η Κομισιόν. Το είπα και στην προηγούμενη συζήτηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Κομισιόν ότι άλλαξαν οι όροι. Να αλλάξει και η κουλτούρα της ιδιαθεσμική της Κομισιόν. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά να παρακολουθήσει ο κύριος ε, Επίτροπος Διεθνούς Εμπορίου και την ταινία, μια παλιότερη ταινία, The Negotiator, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θα μάθουν πώς εκπροσωπούν και τα ευρωπαϊκά αγροτικά συμφέροντα προς τα έξω γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ποια συμφέροντα εκπροσωπούν, προτάσουν στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και όχι τα αγροτικά. Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να υπερασπίζουμε το συμφέρον των Ευρωπαίων αγροτών. Την Ευρώπη της υπαίθρου. Κύριε Πρόεδρε, ε, συγκράτησα τις παρατηρήσεις ότι αν είναι κωδικοποιώ τώρα εάν μια συμφωνία στην παγκόσμια εμπορική κλίμακα είναι προτιμότερη, μια παγκόσμια συμφωνία, επομένω γύρω στι Δόχα ή διμερεί συμφωνίε, βλέπω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων τάσεται υπέρ ε, μια ρύθμιση ε, κάτω από την ομπρέλα του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορίου, πράγματι στο γύρο τη Δόχα. Τώρα αυτό θα έδινε περισσότερη ε, ασφάλεια, θα αποσαφήνιζε ρόλου, καταστάσει αλλά και εδώ όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει ήδη από τον Οκτώβριο του 2005 μια πάρα πολύ γενναιόδορη προσφορά δεν ανταποκρίθηκαν άλλοι εταίροι, δεν ανταποκρίθηκαν ανταγωνιστικές δυνάμεις σε αυτή την προσφορά. Συγκράτησα, ε, και εύχομαι και εγώ να, να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις προς ε, αλλά όπως πολύ σωστά είπαν και οι συνάδελφοι, μιλούμε για, ένα, για μια ισόρροπη συμφωνία για να fair, όπως λέγεται και στην διάλεκτο, ε, ε, εμπορικό σύστημα, ε, για ένα ισόρροπο εμπορικό σύστημα, για ένα δίκαιο εμπορικό σύστημα και δεν μπορούμε να βάζουμε σε αυτές τις παραχωρήσεις στην ίδια μοίρα της χώρας της Αφρικής, όπως αναφέρθηκε εδώ, με τις, ανα... ανταγωνίστριες δυνάμεις, οι οποίοι είναι εξ... και ανταγωνίζονται με αθέμητους όρους την ε, ευρωπαϊκή γεωργία. Και για την Αφρική πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες, το Everything But Arms, υπάρχει ε, όλα πλην όπλων, υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς έχει απονημηθεί στην Αφρική, ε, δεν το έχουν κάνει όμως άλλοι εταίροι στο πλαίσιο του παγκοσμίου εμπορίου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκράτησα τις παρατηρήσεις ότι να μην υπάρχουν κακές διαπραγματεύσεις, ε, επομένως κακές παραχωρήσεις. Δεν είναι η λύση οι αποζημιώσεις. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα ε, με αυτή την παρατήρηση. Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι γεωργοί στην παραγωγή τους. Και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να δίνουμε αποζημιώσεις, αποζημιώσεις για την, ε, θέματα τώρα το animal welfare και νομίζω ότι εξαντλήθηκε και βρέθηκε και μια τομή. Εγώ ανήκω σε αυτούς που λέω ότι κοιτάξτε έχουμε το animal welfare ε, να είναι κοινή πολιτική, αγροτική, αλλά η δημόσια υγεία για τους ανθρώπους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία μόνο συντονιστική αρμοδιότητα. Ως γνωστόν η δημόσια υγεία ως ευρωπαϊκή πολιτική είναι συντονιστική ε, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έτσι ήθελαν τα κυρίαρχα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ με την, ε, απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Μαγκίνες, για την, ε, στην τροπολογία 38 για το impact, ε, την ανάγκη impact ε, assessment. Ε, μπορώ να κάνω και άλλες παρατηρήσεις, αλλά νομίζω κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, αυτό που ήθελα να πω είναι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την Κομισιόν βεβαίως για, τις, για τη συνεισφορά τους, για τις τροπολογίες και νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα που θα κωδικοποιεί κατά τρόπο αρμονικό αλλά και δίκαιο ε, και ζωντανό τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο ε, είναι ευρωπαϊκό αλλά ε, αγγίζει και τα διεθνή όρια της Ευρωπα... την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πάπαγαμ Στάμκο και να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους που πήραν το λόγο. Τελειώνουμε εδώ. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στις 3, το υπενθυμίζω, με την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά από το 2013. Αλμπερτές και ο διευθυντή επίσης τάσο Ανιώτης από τη Γενική Δεύση Γεωργίας θα είναι παρόν. Λοιπόν, πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της ΚΑΠ. Στις 3 εδώ. Γεια σας και καλό γεύμα.